Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ε, η εξέταση θα γίνει στο 12, η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η επόμενη σημεία είναι Δημοσιονομικός Λόγος Ανθρωπιστικής Βοήθειας του, του κυρίου Χάουζα. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι μεγαλύτεροι δότε της ανθρωπικής βοήθειας. Η Γενική Διευθυνσή ΕΚΟ διαχειρίζεται ένα τεράστιο ποσοστό, 1,1 δις δηλαδή ευρώ το περασμένο έτος. Έχω παίζει ένα ρόλο συντονισμού και η εφαρμογή επιτόπου θα γίνεται πάντα από διάφορους εταίρους μας, δηλαδή μη κυβερνήσεις οργανώσεις, ε, υπηρεσίες του ΟΗΕ, αλλά και άλλες διεθνείς οργανώσεις είναι γεγονός ότι με την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή βοηθούνται εκείνοι που έχουν περισσότερες ανάγκες στον κόσμο και εάν δεν είμαστε αποτελεσματικοί έχουμε ε, ανθρώπινα θύματα. Και γι' αυτό είναι καλό που το Κοινοβούλιο εξετάζει μετά από κάποια χρόνια την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και της εφαρμογής το αποτέλεσμα είναι ότι όσον αφορά η, τη συνεργασία μεταξύ της έχω και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το πρόγραμμα αυτό, έχω να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ε, συλλογές και καλή συνεργασία μεταξύ Γενικής Διευθυντής ΕΚΟ και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης, το 2008 η Συμφωνία Πλαίσιο οδήγησε σε πρόοδο υπάρχει μια αναθεώρηση αυτή τη χρονιά και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διακατεύθυνση. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ε, της μείωσης του γραφειοκρατικού κόστους. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον ΟΗΕ, το θέμα είναι κάπως κρίσιμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κοινοτική μέθοδος τη εφαρμογή του προπολογισμού ε, έχει κάποια προβλήματα όσον αφορά τον αποτελεσματικό ε, έλεγχο της αποτελεσματικότητα ε, χρήση των πόρων αυτών. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή, αυτός ο ενιαίος έλεγχος. Καταρχήν να υπάρχει πρόσβαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια έκθεση ελέγχου των λογιστικών του ΟΕΕ και νομίζω ότι γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του για τον έλεγχο. Επίση, οι επιμέρου εκθέσει που υποβάλλονται στην Κομισιόν όσον αφορά την εφαρμογή, κατά τη γνώμη μου, ε, δεν είναι σωστά διατυπωμένε. Θα πρέπει να έχουν πιο πολύ ουσία στο περιεχόμενο, να μην είναι τόσο ασαφή, Επίση, ε, θα πρέπει να κάνουμε του ελέγχου μετά το σκάνδαλο αυτό με την βορειοκορεϊκή κυβέρνηση, να δούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόοδος και εδώ καλούνται βέβαια τα κρατη να ασκήσουν πίωση στα Ηνωμένα Έθνη. Όσον αφορά την εφαρμογή, με τις μη κυβερνικέ οργανώσει υπάρχουν κάποια δύναμα σημεία, ιδίως όσον αφορά, όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης κάποιες μη κυβερνικές οργανώσεις, γιατί πολλές φορές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν έχουν τις απαραίτητες δομές. Επίσης, όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου, υπάρχουν ελλείψεις. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι άλλοι εταίροι μας να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την διαχείριση των πόρων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί εσωτερικών ελέγχων. Όσον αφορά το κόστος υποστήριξης, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ένα τρίτο σημείο, υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ σε παρόμοια προγράμματα και θα ήταν καλό να έχουμε ενιαία σημεία προσδορισμού για παρόμοια προγράμματα για να αποφύγουμε την μη αποτελεσματική χρήση. Στο μέλλον είναι επίσης σημαντικό να συζητάμε για την ε, αηφορία και την πρόληψη, παραδείγματος όσον αφορά την πρόληψη καταστροφών με τη δημιουργία συστημάτων έγκρισης προειδοποίησης, επίσης ανθρωπιστική βοήθεια για αναπτυξιακή βοήθεια, να βελτιώσουμε και αυτό το τομέα και επίσης θα πρέπει να δώσουμε καλές δυνατότητες στον τοπικό πληθυσμό αναπτύσσοντας τις ε, απαραίτητες τοπικές δομές. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι έρχεται αυτή και στην αρμόδια επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία και θα χαρώ να τύχει η πλειοψηφία και στην Ολομερή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ, συνάδελφε Ερνχάου. Σα περνάμε στη διαδικασία Κάτσου και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ρούμπικ. Κυρίε και κύριοι, έχουμε εδώ με την έκθεση αυτή δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει μεγάλη ευθύνη στην ανάπτυξη και τα μέτρα βοήθεια τα οποία προσφέρουμε πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να φτάνουν πράγματι στον κόσμο, στους ανθρώπους που πράγματι τα χρειάζονται και να φέρουν αποτελέσματα. Αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέσουμε και ενέργεια στις πιο, φτωχές, στις πιο περιοχές, μέτρα δηλαδή αναπτυξιακά τα οποία θα εξασφαλίσουν και τις ε, ενεργειακές ανάγκες του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε, να διαμορφώσουμε κατά τρόπο αιφόρο τους σπόρους. Χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις πιστεύω στο κείμενο και θα πρέπει ως εκ τούτου να εργαστούμε έτσι ώστε να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο μακροπρόθεσμα, βιώσιμα δηλαδή, θα μας επιτρέψει την υλοποίηση των αναπτυξιακών μας στόχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούμπιχ, κυρία Τίτσα. Τσίκαο. Ευχαριστώ. Δεδομένης της ε, αύξησης, της συχνότητας, της σοβαρότητας των ανθρωπιστικών καταστροφών που πλήττουν πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής προκειμένου να αυξηθεί ο προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια από το 2014 με μια αύξηση 915 εκατομμυρίων το χρόνο. Επίσης το αποθεματικό έχει αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια για την ίδια περίοδο. Και υπάρχει επίσης και η πρόταση του χρόνου να χρησιμοποιηθούν όσα χρήματα βρίσκονται στο αποθεματικό και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να φροντίσουμε για την πρόληψη και για την άμεση αντιμετώπιση καταστροφών εφόσον αυτές προκύπτουν. Εμείς πιστεύουμε ότι τα παιδιά οι έγκυοι, οι γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά πρέπει να υποφελούνται κατά προτεραιότητα από την χορήγηση ιατρικών ε, υπηρεσιών και τροφίμων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τσικά. Κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ένας όρος ε, για ένα προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημοσιονομικών ελέγχων αλλά και της αναπτυξιακής βοήθειας είναι η αξιολόγηση των αναγκών σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Πολλά μπορούμε να κάνουμε όπως βλέπουμε στο κέρας της Αφρικής παρά την εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια δεν υπάρχει καμία επιτυχία εκεί. Πολλοί πόροι φτάνουν εκεί, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι τους παίρνουν. Είναι απαραίτητο να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια ώστε να μπορούμε να ε, εντοπίσουμε τους ε, παραλήπτες των ενίσχυτων της βοήθειας και να μπορούμε να τους ε, βρούμε. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στην έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εστιάσει την προσοχή στον έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και στη συνεργασία με, άλλες, με άλλους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματά της για ανθρωπιστική βοήθεια έχουν ως στόχο να ανακουφίζουν τα θύματα καταστροφών, φυσικών καταστροφών ή θύματα πολέμου και είναι μια πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες αυτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζεται με πάνω από 200 οργανώσεις που ακολουθούν όμως πολλές και διαφορετικές στρατηγικές η καθεμία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σημαντικούς πόρους που έχουν ως στόχο την ανακούφιση των θυμάτων. Όμως, οι μηχανισμοί ελέγχου είναι επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή της ε, δίκησης ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι γι' αυτό και θεωρώ ότι πρώτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που βελτιώνει και τον έλεγχο των δαπανών στον τομέα αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό και έχει ως στόχο καλύτερη ποιότητα στις δαπάνες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ. Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών ανά τον κόσμο. Ταυτόχρονα ο προπολογισμό της Ένωσης που προορίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία των διαρκώς περικόπτεται. Ως προς αυτό χρειάζεται σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η Ένωση χρειάζεται ένα ταμείο ανθρωπιστικό πιο ρεαλιστικό. Υπογραμμίζω την ανάγκη να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στη χρηματοδότηση των ενεργειών για πρόληψη των καταστροφών και της επίγουσας βοήθειας. Είναι απαραίτητο η Ευρώπη να έχει ε, επίσημους μηχανισμούς για να μπορεί να προλαμβάνει πιθανούς, πιθανές καταχρήσεις. Ε, η διαφάνεια της συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς είναι λοιπόν πολύ σημαντική. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνοχή ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή. Αντί, αν όχι, Μπορεί αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, η υπερβολική επισητιστική βοήθεια μπορεί να αποθαρρύνει την τοπική παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσα προέκυψαν σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από πλευρά τη Κομισιόν, ε, γιατί υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί το ανθρωπιστικό ταμείο, να ενισχυθεί <clears throat> αυτή η δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι αναγκαιότητα ο διαχωρισμό το είπε μόλις η συνάδελφο Μπασέσκου, πολύ κέρια, ότι πρέπει να διαχωριστεί η πρόληψη από την επίγουσα βοήθεια. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, αναγκαιότητα να υπάρξουν πιο διαφανείς μηχανισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων. Πριν από κάποιες εβδομάδες υπέβαλα μια ερώτηση για μια υπόθεση που προέκυψε και βγήκε στις ε, εφημερίδες ολόκληρη της Ιταλίας ενός άνεργου νέου που ασχολείται σε μια ΜΚΟ που προσπαθούσε να ζητεί χρήματα χωρί κανένα σύμβαση, χωρίς κανένα συμβόλο εργασίας. Τι κάνουν οι άνεργοι λοιπόν, κάνουν τους κυνηγού επιδοτήσεων για τις ΜΚΟ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερος έλεγχος σε διαφάνεια σε αυτών των μηχανισμών και δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλβέστρης. Και για να ολοκληρώσουμε εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο θα λάβει η κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή και το προσωπικό εδώ στις Βρυξέλλες που ασχολείται με τα ανθρωπιστικά ζητήματα που βοηθούν πάνω από 40 χώρες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από ανθρωπιστικές ε, ζημιές που έχουν υποστεί. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά πρέπει να το πω και να ξέρουμε ότι όντω δαπανώνται καλά τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ζούμε σε καιρού όπου έχουμε όλο και περισσότερες καταστροφές. Δεν έχουμε όμως όλο και περισσότερα χρήματα, κάτι το οποίο μας πιέζει ακόμα περισσότερο για το πώς δαπανάμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, για το πώς δουλεύουμε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν Είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, συμβουλές που μας δίνετε. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία. Πρώτον, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή που έρχεται η έκθεση αυτή. Και αυτό γιατί δουλεύουμε πάνω στην αναθεώρηση της ε, συμφωνίας μας εταιρικής σχέσης και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για καλούς ελέγχους, για καλά συστήματα ελέγχων που να είναι και ταχύτητα. Βλέπετε, η ταχύτητα για μας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Σημαίνει ότι σώζονται ζωές και σημαίνει ότι θα πανάμε και λιγότερα χρήματα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα Ηνωμένα Έθνη. Πολύ ορθά λέτε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να έχουμε διαπραγματεύσεις προκειμένου η εσωτερική έλεγχη να διατίθεται και σε μας. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ελέγχουμε την ε, ποιότητα των ε, προσπαθειών, των προγραμμάτων των ε, εταίρων μας. Κατά πόσο ανταποκρίνονται δηλαδή στα υψηλέ ε, προδιαγραφές που έχουμε θέσει εμείς. Υπογραμμίσουμε επίσης και στις διάφορες εταιρικέ συμφωνίες που συνυπογράφουμε το θέμα των αποτελεσμάτων. Ναι, 1,1 δις ευρώ δαπανάμε ανά τον κόσμο για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους, όντως. Έχουμε φτάσει στα 146 εκατομμύρια θύματα όμως, τα οποία δίνουμε τρόφιμα, ε, θέρμανση, ένα, μια σκεπή κάτω από την οποία να μπορούν να ζήσουν. Δυστυχώς οι κίνδυνοι αυξάνονται, η αστάθεια να το κόσμο αυξάνεται. Γι' αυτό και οι εταίροι μας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν για να πιάνουν τόπο τα χρήματά μας. Τέλος, συμφωνώ απόλυτα με τη σύστασή σας όσον αφορά την ε, ανακούφιση και τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τις δαπάνες μας για ανθρωπιστική βοήθεια, έχοντας όμως βέβαια πάντα καλά αποτελέσματα. Πώς θα προλαμβάνουμε δηλαδή τις καταστροφές και πώς θα μειώνονται τα καταστροφικά αποτελέσματα από αυτές. Και όλα αυτά τα κάνουμε και σε συνεργασία με τον Επίτροπο Αμπίλγας. Βλέπετε, ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε είναι η επιμονή και η ανάπτυξη. Στο έργο μας θέλουμε να συμπεριλάβουμε μία συστηματική ανάλυση κόστους-οφέλους έτσι ώστε να μπορούμε να προτείνουμε προγράμματα και σχέδια τα οποία να ανταποκρίνονται στους στόχους μας που είναι τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι σε εμά έχετε και θα βρίσκετε πάντα έναν πολύ καλό εταίρο, ο οποίος θέλει να βοηθήσει για την ανακούφιση του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γεωργίεβα. Έληξε η συζήτηση για αυτό το θέμα και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 12. Οπότε διακόπτουμε μέχρι τότε.